το άδικη πρόταση ανεξάρτητα από τα αριθμητικά στοιχεία ε, που προβλέπει το πολιετές. Γιατί ε, δεν επιτρέπεται να δημιουργούνται ομάδες πλούσιων και φτωχών κρατών ή να ε, υποβαθμίζεται το επίπεδο. Θα πρέπει να δούμε και τα στοιχεία του προϋπολογισμού. Ας δούμε τα αριθμητικά στοιχεία του προϋπολογισμού. Ας δούμε την διαφορά μεταξύ του υψη, της υψηλότερης και της χαμηλότερης πρότασης. Αυτά είναι 350 εκατομμύρια. Αυτό σημαίνει ανά ε, μήνα, ανά πολίτη, 9 ευρώ. Αυτή είναι η διαφορά. 9 ευρώ διαφορά ανά πολίτη θα είναι ακριβό έτσι το μέλλον της Ευρώπης. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Πρόεδρε, εξότιμοι συνάδελφοι, στις τελευταίες ε, διαπραγματεύσεις για το πολιτερές δημοσιονομικό πλαίσιο στις 8 ε, Φεβρουαρίου 2013 πέτυχαν μια συμφωνία η προηγούμενη ήταν το 2012. Την υπόλοιπη ιστορία την γνωρίζουμε. Επίσημα αποφασίστηκε στις 2 Δεκεμβρίου 2013 στη συνέχεια ε, μέσω της χρηματοδότησης πολλά προγράμματα έπρεπε να βρουν άλλες χρηματοδοτικές ε, πηγές. Ε, δικαιολογημένα είπε τότε ο κύριος Ερτιγκερ ότι δεν υπήρχαν καθόλου πόροι, καθόλου ποστά απορρόφησης. Ε, ε, εμείς είμαστε στο δρόμο να κάνουμε το 2020 πάλι ένα χαμένο χρόνο προς τον προπολογισμό. Μετά το Brexit ε, και το αίτημα της ε, βιωσιμότητας, τι κάνουμε, της βιώσιμης ανάπτυξης. Όλοι όσοι, όλες όσες χώρες κοιτάνε το δικό τους προπολογισμό προσκαλούνται θερμά να δουν τις προτάσεις του σώματος για ένα καλύτερο σύστημα ιδίων πόρων. Ε, μόνο έτσι θα μπορέσουμε να είμαστε αποφασιστικοί να λύσουμε τα κοινά προβλήματα στις 20 Φεβρουαρίου. Ο κύριος... Χάβα, παρακαλώ. Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να έχει πρόσβαση στα κονδύλια του επόμενου πουδουπού το συντομότερο δυνατό με τον πιο προκλέψιμο τρόπο. Έχουμε μία συνεισφορά για τα, των κρατών μελών για την επόμενη περίοδο προγραμματισμού. Μιλάμε για ένα ευρώ που επενδύεται έχουμε 9 ευρώ που επιστρέφονται στη χώρα μας. Σούπερ. Οι υπηρεσίες της Κομισιόν λένε ότι υπάρχουν προβλήματα. Η Φιλανδία θα συνεισφέρει 22 δισεκατομμύρια ευρώ και θα πάρει 13,2 δισεκατομμύρια πίσω. Εμείς θα, σε εμάς θα επιστραφούν 16,5 δισεκατομμύρια στην Ρουμανία. Εμείς θέλουμε κονδύλια για επενδύσεις, για να καταπολεμήσουμε τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα πρέπει να βρεθεί σύντομα μια πολιτική συμφωνία. Thank you. Mr. Tang, for one minute. Ο κύριος Τάγκ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα μιλήσω Ολλανδικά. Αν διαβάζετε τις εφημερίες, θα βλέπετε ότι μία φορά τα 7 χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μια τεράστια ευκαιρία για να βρει τις κατάλληλες απαντήσεις στις προκλήσεις. Να βελτιώσει τις ισοδομικές συνδέσεις στην Ευρώπη. Να προωθήσει την ευρωπαϊκή επιστήμη. Όμως, οι εφημερίδες δεν μιλάνε καθόλου για το κόστος του προϋπολογισμού. Καταρχάς λοιπόν, δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στις ε, μεγάλες ε, επιχειρήσεις να μην πληρώνουν το κόστος της εσωτερικής αγοράς. Ούτε μπορούμε να ε, κολλάμε στο 0,001% δεν πρέπει να κοιτάμε τα ποσοστά. Θα πρέπει να επιλέγουμε τις ευκαιρίες. Θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε με τα δεδομένα μας. Ο κύριος Χαρά, σε ένα λεπτό. Ε, κυρία Πρόεδρε, κύριε, Επίτροπε, εγώ ε, ζητώ ειλικρίνεια στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό. Αφορά το μέλλον μας και Γι' αυτό κάνει ενημερωτική εκστρατεία το Κοινοβούλιο, γιατί οι πολίτες κατά πλειοψηφία πιστεύουν ότι τα πιο πολλά κονδύλια ε, πηγαίνουν στην διοίκηση, ενώ το 94% των κονδυλίων ε, δίνονται στις περιφέρειες για την Ήπεθρο, για τα πανεπιστήμια, τις επιχειρήσεις, την ανάπτυξη, ε, την επένδυση στο μέλλον. Κάθε ευρώ ε, ε, ε, δημιουργεί 3 ευρώ στις χώρες. Αποσιωπάται η προστιθέμενη αξία η οποία είναι πολύ μεγαλύτερη από ό,τι συνεισφορά. Δεν υπάρχουν καθαροί συνεισφέροντες διότι τα έργα, η αξία που δημιουργείται και παράγεται ε, ξεπερνάει πολύ την εισφορά. Είναι λοιπόν λάθος να το λέμε αυτό. Πού είναι οι μεγαλύτερες διαφορές στην παιδεία, την έρευνα, στις επενδύσεις, στο Green Deal, στην ανάπτυξη της υπαίθρου, την ασφάλεια, την κοινωνική συνοχή. Ε, ε, ε κύριε Επίτροπε, κυρία Προεδρεύουσα στο Συμβούλιο, θα πρέπει να φροντίσουμε ε, για το καλό των πολιτών και ε, να κλείσουμε το κενό του προϋπολογισμού με ένα, μια σωστή προσέγγιση στο σύστημα των ιδίων πόρων. Κύριε Κάρας, υπάρχει μπλε κάρτα του κυρίου Νεγκρέσκου. Δέχεστε την ερώτηση, κύριε Κάρας. Α, όχι, όχι, όχι. Α, όχι, όχι, όχι, δεν ζητήθηκε. Ε, ε, ε, <laughs> κύριε Κάρα, δεν υπάρχει πρόβλημα, δεν ζητήθηκε ε, μπλε κάρτα. Τελευταίος ομιλητή στον του μου είναι ο κύριος Μεϊμαράκης. Ένα λεπτό, παρακαλώ. Τα επόμενα χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση καλείται να υλοποιήσει το Green Deal, μια εξαιρετικά φιλόδοξη πολιτική. Και η επιτυχία αυτής της πολιτικής θα κρεθεί από την ικανότητά μας ως νομοθέτες να εξασφαλίσουμε την ίση μετάβαση των κοινωνιών μας στην πράσινη οικονομία και για να μπορέσει αυτό να υλοποιηθεί χωρίς ανισότητες δεν επαρκεί η συνεισφορά του 1% από τους ετήσιους εθνικούς προϋπολογισμούς. μέχρι τώρα με το ποσό αυτό η ευρωπαϊκή ένωση υλοποιούσε πολιτικές ορόσημα όπως ήταν η κοινή αγροτική πολιτική και η πολιτική συνοχής. και θέλουν κάποιοι με την ίδια χρηματοδότηση να εφαρμόσει και την πιο φιλόδοξη πολιτική των τελευταίων ετών. ε αυτό δεν γίνεται. νέες πολιτικές απαιτούν νέες χρηματοδοτήσεις. η πρόταση λοιπόν του κοινοβουλίου για ένα τρία θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ λογική και εξασφαλίζει την υλοποίηση των πολιτικών που δικαιώνει τα οράματα των πολιτών για την ευρώπη του μέλλοντος. χωρίς να περικόπτει τις απαραίτητες χρηματοδοτήσεις για την υλοποίηση της αγροτικής πολιτικής και της πολιτικής συνοχής και μπορεί ταυτόχρονα με τη μεγαλύτερη χρηματοδότηση να εξυπηρετηθούν όλες αυτές οι ανάγκες. γι' αυτό και δεν είναι υπεύθυνο να γίνονται βαρισίμαντες εξαγγελίες από τις εθνικές κυβερνήσεις χωρίς αυτές να συνοδεύονται από τολμηρές πρωτοβουλίες και χρηματοδότηση. η πρόταση του κοινοβουλίου περιμένουμε και πρέπει να γίνει αποδεκτή. ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Πάμε τώρα στη διαδικασία Catch the Eye. Πρώτος, ε, η, κυρία Μοντινέρο Τάγκυλα, πρώτη ομιλήτρια. <clears throat> Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η θέση μας εδώ στο Κοινοβούλιο είναι ξεκάθαρη πλέον. Δεν συμφωνούμε με λιγότερα κονδύλια, στο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο και θα Αυτό που ζητάμε είναι σημαντικό για την οικονομική ανάπτυξη των χωρών μας. Δεν συμφωνούμε με περικοπές σε βάρος των χωρών και της χώρας μου της Πορτογαλίας. Χρειαζόμαστε μια πολιτική η οποία ε, θα ανταποκρίνεται με τον τρόπο που πρέπει στην ΚΑΠ και την πολιτική συνοχής. Πολύ σημαντικά και τα δύο για τη χώρα μου. Υπάρχουν πολλές επιφυλάξεις, ανησυχίες ε, από πολλές χώρες, Πορτογαλία, Ισπανία, Γαλλία, διότι ε, έχουν ε, προβληματικές περιοχές που πρέπει και αυτές να έχουν τη δυνατότητα να αναπτυχθούν. Υπάρχουν και προβλήματα αλληλείας, προβλήματα οικονομικά, προβλήματα που αφορούν τον τουρισμό και όλα αυτά δεν θα πρέπει να ε, υποβαθμιστούν. Χρειαζόμαστε μια ένωση για τους περιφέρειες και ένα προϋπολογισμό χωρίς περικοπές. Επόμενη, επόμενος ομιλητής είναι ο κύριος Νεγκρέσκου. Ε, εδώ και δύο χρόνια για πρώτη φορά είχαμε μια συνθήκη ε, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για τον προπολογισμό. Έκτοτε δεν βρέθηκε καμία λύση. Ίσως ήρθε κατάλληλη στιγμή για να σκεφτούμε την Ευρώπη του αύριο. Έχουμε ανάγκη έναν επαρκή προπολογισμό και ανώτερε συνεισφορέ εκ μέρου των χωρών μελών. Ε, ε δεν υπάρχουν ναι, προτεραιότητες. Η μόνη μας προτεραιότητα είναι ο Ευρωπαίος πολίτης. Άρα έχουμε ένα ανάγκη ένα προπολογισμό ο οποίος θέλει κονδύλια για την γεωργία, για το περιβάλλον, για την εκπαίδευση κλπ. Εφόσον είμαστε διατεθειμένοι να πάρουμε αποφάσεις σήμερα μπορούμε να το κάνουμε. Άρα το Συμβούλιο θα πρέπει να πάρει μία απόφαση. Έχουν υποβληθεί προτάσεις, θα πρέπει να σταθεί στο ύψος της ευθύνης του το Συμβούλιο προκειμένου να προχωρήσουμε. Οι Ευρωπαίοι πολίτες πολίτες έχουν ε, υψηλές προσδοκίες απέναντί μας προκειμένου να υποστηρίξουμε αυτόν τον προϋπολογισμό. Η κυρία Γουίλα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Αυτή η συζήτηση στην Ολομέλεια έδειξε τρεις ε, μεγάλες συμπτώσεις στο ε, περιθώριο των αποκλήσεων. Όλοι έχουμε γνώση των ε, δυσκολιών που προποθέτει η κατάρτιση του προπολογισμού στο πλαίσιο του Brexit. Γι' αυτό είμαστε υπέρ μια ταχεία συμφωνία η οποία θα παρέχει νομική ασφάλεια στου βασικού τομεί τη οικονομία μα. Ζητούμε επίση ε, πέρα από τους αριθμούς, ένα προπολογισμό που ανταποκρίνεται στις νέες προτεραιότητες. Το Green Deal θα είναι η προτεραιότητά μας, αλλά αυτό, αυτή η συμφωνία και όλες ε, οι πρωτοβουλίες, όπως για παράδειγμα ε, όλες οι πρωτοβουλίες θα πρέπει ε, να έχουν τη συνένεση των Ευρωπαίων πολιτών. Ε, θα πρέπει όμως να δώσουμε και στους γεωργούς την αναγκαία υποστήριξη, όχι μόνο για να εκπληρώσουν πιο φιλόδοξους οικολογικούς στόχους, αλλά για να έχουν και μια οικονομική δραστηριότητα που να τους αποδίδει. Θα πρέπει να πάψουμε, να δώσουμε ένα τέλος στις ματαιώσεις των γεωργών μας. Ε, γιατί είναι μεγάλες οι προκλήσεις για την Ήπεθρο και είναι σημαντική η συνεισφορά της στη βιωσιμότητα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ο κύριος Γόλας. Ε, ε, κυρία Πρόεδρε, αν η Ένωση θέλει να χρηματοδοτήσει όπως πρέπει το Ιμπράσιν Συμφωνία, την ΚΑΠ, τη συνοχή και να διατηρήσει και την ειρήνη, θα πρέπει να ε, αξιοποιήσουμε την ευκαιρία του Brexit και να αποφύγουμε και την άσκοπη στρατιωτικοποίηση της Ευρώπης. Ε, να αποφύγουμε μέτρα και άλλα μέτρα που ε, προτάθηκαν από ανθρώπους που είναι υπό τον έλεγχο των, της στρατιωτικής βιομηχανίας. Επίσης, θα πρέπει να κινηθούμε προς τα καθαρά τρόφιμα, χωρίς ε, ε, επικίνδυνα, ε, επικίνδυνες ουσίες, ζυζανιοκτώνα κλπ. Θα πρέπει να βοηθήσουμε τους αγρότες να επιβιώσουν παράγοντας ταυτόχρονα πιο καθαρά τρόφιμα. Δεν χρειαζόμαστε μεγαλύτερο προϋπολογισμό. Πρέπει όμως να είναι καλύτερος. Δεν είναι αποδεκτό ε, να αυξάνουμε τον προϋπολογισμό σε βάρος των πολιτών της Ευρώπης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ε, θα πρέπει να προχωρήσουμε με τρόπο ορθολογικό. Θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο... Ε, ε ρεαλιστές ε, να διατηρήσουμε αυτά τα έργα που είναι καλά και είναι αρκετά. Ε, ε, εμείς από κοινού μπορούμε να κάνουμε περισσότερα πράγματα και για το κλίμα και για την ασφάλεια, την έρευνα, τις επιστήμες, τις νέες τεχνολογίες, την έρευνα για τον καρκίνο κλπ. Υπάρχουν έργα που αφορούν τον άνθρωπο ε, πάντα πρέπει να έχουμε υπόψη μας τις κοινέ μας αξίες, γιατί είμαστε μαζί. Οι καθαροί χρηματοδότες δεν πρέπει να ξεχνούν την αλληλεγγύη, ούτε πρέπει να ξεχνούν ότι ε, ωφελούνται αν δώσουν ε, χρήματα ε, σε φτωχότερες χώρες. Αυξάνονται οι εξαγωγές αυτοκινήτων τους, αυξάνονται, αυξάνεται η παραγωγή τους και τα ωφέλη τους. Πολλές φορές ε, οι ευρωπαϊκοί κανόνες δεν τηρούνται. Δεν πρέπει να ξεχνάμε το μέλλον, γι' αυτό πρέπει να έχουμε και τον ανάλογο προϋπολογισμό. κυρία Καράρες. κυρία Καρβάλιες, έχετε το λόγο. Χωρίς μικρόφωνο. Μερικέ φορέ και εγώ δεν καταλαβαίνω το όνομά μου. Επιτρέπετε να κάνετε λάθη. Εγώ φταίω, λέει η Πρόεδρος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αυτά που θα σας πω ακούστηκαν και από άλλους, αλλά αισθάνομαι υποχρεωμένη να, το, να τα πω και εγώ για διοντολογικούς λόγους. Η Κομισιόν μας παρουσιάζει ένα πρόγραμμα εργασίας πάρα πολύ φιλόδοξο για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις της Ευρώπης μας. Θα πρέπει όμως σε αυτή την ε, ε, απάντηση που δίνουμε να μην υπάρχουν θυσίες, να μην θυσιάζουμε τις πολιτικές που διαρθρώνουν και διαμορφώνουν τις ε, κοινωνίες μας. Δεν πρέπει να υπάρχει μια διχοτόμηση ανάμεσα στις παραδοσιακές και στις μοντέρνες πολιτικές. Και εδώ μιλάω συγκεκριμένα για την ανάγκη να διατηρήσουμε, να ενισχύσουμε την πρικοδότηση του προπολογισμού για σημαντικέ ε, πολιτικέ όπω η κοινή γεωργική πολιτική, η αληθική πολιτική, η περιφερειακή πολιτική. Γιατί αν δεν το κάνουμε, οι πολίτε μα δεν θα καταλάβουν τι νόημα έχει και πού κατευθύνεται η ευρωπαϊκή οικοδόμηση. Κάνω αυτή την έκκληση, ούτως ώστε αυτέ οι διαρθρωτικές πολιτικές, οι βασικές πολιτικές, να συνεχίσουν και να επενδύσει σε αυτές και στο μέλλον η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ο κ. Πεκοράινεν, για ένα λεπτό. Θα προσπαθήσω ξανά. Μπορεί να, το λέω, να το λέω λάθος το όνομα. Ο κύριος Πεκοράινεν. Είστε εδώ. Arvoisa, arvoisa puheenjohtaja, ναι, εδώ είμαι, Πρόεδρε. Μάλιστα. Τι μήνυμα περνάει από αυτή τη συζήτηση. 1,7%. Τι είναι αυτό. Αρκεί αυτός ο προϋπολογισμός. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να κοιτάξουμε τις προτεραιότητες και πού ξοδεύονται τα χρήματα. Επίσης, ε, πώς ε, κατανέμονται τα καθήκοντα ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα κράτη-μέλη. Σε ορισμένου τομεί, τα κράτη-μέλη πρέπει να έχουν περισσότερε αρμοδιότητε. Παραδείγματο χάρη, στο πώ θα μειώσουν τι ανισότητε σε εθνικό επίπεδο. Καθώ θα μειωθούν, πώ θα μειωθούν οι ανισότητε μεταξύ των χωρών. Οι ανισότητε αυτέ δεν έχουν μειωθεί. μειωθεί. Θα πρέπει τα λεφτά τη Ευρωπαϊκή Ένωση και τα εθνικά κονδύλια να χρησιμοποιούνται με τέτοιο τρόπο, ούτω ώστε να υπάρχει και μια σωστή ισορροπία μεταξύ των διαφορών περιφερειών ή τη χρηματοδότηση, τη έρευνα και τη ανάπτυξη. Υπάρχουν πολλές ευθύνες των κρατών μελών. Πολλές επενδύσεις στην εκπαίδευση, στην έρευνα και στην ανάπτυξη σε ορισμένε χώρες είναι πάρα πολύ μικρές. Αν θέλουν να δώσουν προτεραιότητα κάποιε χώρες σε αυτό το τομέα, στη χώρα τους ας πούμε, ας το κάνουν. Αυτό έχει απόλυτο νόημα. Ο κύριος Χριστοφόρου. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πιστεύω ότι οφείλουμε να είμαστε ειλικρινεί και με τους εαυτούς μας και προς τους Ευρωπαίους πολίτες. Εάν είμαστε πραγματικοί ευρωπαϊστές, εάν πραγματικά θέλουμε και διεκδικούμε μια καλύτερη και μια πιο ισχυρή Ευρώπη, εάν θέλουμε πραγματικά η ευρώπη να έχει μέλλον και προοπτική και να μπορέσει να χρηματοδοτήσει τα μεγάλα οράματα και φιλοδοξίε τη όπω είναι η πράσινη πολιτική η καταπολέμηση του καρκίνου ο ευρωπαϊκό στρατό η γενιαία αμυντική άμυνα και ασφάλεια τότε ένα τρόπο υπάρχει μια προπόθετη προπόθεση να επαυξηθεί ο προπολογισμό από το 1 τη συνεισφορά των χωρών μελών στο 1,3 δεν μπορεί διαφορετικά να έχουμε μεγάλες φιλοδοξίες μεγάλα οράματα και μεγάλα λόγια δεν μπορούν να χωρέσουν σε έναν προπολογισμό όπου τα κράτη συνεισφέρουν μόνο ένα εγώ στηρίζω τη θέση και την άποψη του αγαπητού προέδρου της ομάδας μου του Μάφρε Βέπερ ότι δεν μπορούν χώρες οι οποίες δεν εφαρμόζουν το κράτος δικαίου το ευρωπαϊκό και διεθνέ δίκαιο να λαμβάνουν έστω και ένα ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πρώτη και καλύτερη που πρέπει να εξαιρεθεί από αυτά τα κονδύλια είναι η Τουρκία η οποία δεν τα σέβεται και δεν τα εφαρμόζει έτσι λοιπόν τελειώνοντα εάν θέλουμε αυτή η ευρώπη να έχει ισχυρό μέλλον ισχυρή προοπτική και να είμαστε περήφανοι χρειάζεται ένα ισχυρός προϋπολογισμός που να ανταπεκρίνεται στις απαιτήσεις των καιρών. ευχαριστώ. Κύριε Γκραπίνη, ευχαριστώ Πρόεδρε. Επίτροπε, η σημερινή συζήτηση αφορά το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και είναι αξιολύπητο που ο νέος πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου είναι απόν. Θα κάνουμε μια συνεδρίαση για το θέμα αυτό, για τη λάμπη δια της απουσίας του. Ας ε, φτάσουμε όμως στη σημασία αυτού του νέου ε, πουδουπού. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μα είπε ότι θα πρέπει να εξορροπήσουμε τι παλιέ και τι νέε προτεραιότητε. Εγώ πιστεύω ότι οι παλιέ προτεραιότητε εξακολουθούν να είναι επίκαιρε προτεραιότητε. Το... Η κοινή γεωργική πολιτική, η πολιτική συνοχή, δεν μπορούν να απουσιάζουν, ακόμα και αν προσθέσουμε νέες προτεραιότητες όπως ε, η Πράσινη Συμφωνία. Δεν μπορούμε εδώ να βάλουμε στο ίδιο καλάθι την ε, κοινή γεωργική πολιτική με άλλα καινούργια πράγματα και να ξεχάσουμε την πολιτική ας πούμε συνοχής. Ε, επίσης, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι διάφορε επενδύσει που κάνουμε για την ενέργεια και τα λοιπά, τα, υπάρχουν, τα κονδύλια αυτά τα δίνουν οι φορολογούμενοι. Μόνο χάρη στην πολιτική συνοχή όμω θα εξασφαλίσουμε μία Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω τη αλληλεγγύη και μέσω τη κοινή γεωργική πολιτική. Και να προσθέσω κάτι άλλο. Αν έχουμε τι ίδιε επιδοτήσει στη Ρουμανία, στην Τσεχία, στη Γαλλία για του ε, γεωργού, τα ίδια ο Γάλλο και τα ίδια ο Ρουμάνο, δεν μιλάμε για ενιαία αγορά πια. Ο κύριος Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε είναι ότι οι Βρετανοί έφυγαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά η νοοτροπία τους έμεινε πίσω. Αυτά που έλεγε η Θάτσερ, I want my money back, και η αρνητική λογική του Κάμερον, έχουν μεγάλη επιρροή και μετά το Brexit στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, δυστυχώς. Η συνέχιση της Βρετανικής μεθόδου δημιουργεί προβλήματα εμποδίζει την αποτελεσματική λειτουργία της ευρωπαϊκής ένωσης εμποδίζει την αποτελεσματική εφαρμογή των αναγκαίων νέων πολιτικών κυρίως όμως στέλνει ένα μήνυμα παρέτησης σε ό,τι αφορά το κοινό μας ευρωπαϊκό μέλλον. θεωρώ ότι η πρόταση του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου δεν λύνει όλα τα προβλήματα εγγυάται όμως ότι δεν θα ξεφύγουν από τον έλεγχο. ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζουμε για το μέλλον. Ωστόσο, οι νέες προτεραιότητες που έχουν θεσπιστεί δεν σημαίνει ότι οι παλιές προτεραιότητες όπως η συνοχή θα χάσουν τη σημασία τους. Αντιθέτως, οι Ευρωπαίοι περιμένουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση να αυξήσει το επίπεδο διαβίωσης στις περιφέρειες. Γι' αυτό και πρέπει κατά προτεραιότητα να χρηματοδοτηθούν ε, εκείνοι οι στόχοι που έχουν τεθεί, όπως είναι και οι παλιές προτεραιότητες και οι νέες προτεραιότητες. Ο νέος φόρος για τον άνθρακα, η κλιματική αλλαγή. Και όλα αυτά πρέπει να τα συζητήσουμε και να τα παρουσιάσουμε με εύγλωτο τρόπο και ευνόητο τρόπο στους ε, πολίτες μας. Πρέπει να γίνει κατανοητό από τους ανθρώπους στην Ευρώπη ότι ε, όταν ενισχύεται η συνοχή, ενισχύεται και η οικονομία. Ο κύριος Μπασέσκου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σήμερα είχαμε μια συζήτηση που δείχνει πόσο απέχουν οι απόψεις μας. Επιπλέον, διαπιστώνουμε ότι το επίπεδο φιλοδοξιών είναι πολύ διαφορετικό σε σχέση με τα νέα προγράμματα και τις πηγές χρηματοδότησης που όλο ένα και περισσότερο περιορίζονται. Νομίζω ότι βρισκόμαστε σε μια κατάσταση τουλάχιστον παράξενη. Η πιο ορθή λύση θα ήταν τόσο το Συμβούλιο όσο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβουν σοβαρά υπόψη την τοποθέτηση του Ευρωκοινοβουλίου. Δηλαδή 1,3% χρηματοδότηση ώστε να μπορέσουμε να διατηρήσουμε ανέπαθα τα προγράμματα συνοχής, την κοινή αγροτική πολιτική και να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε και να ελοπίσουμε τα νέα προγράμματα που είναι ιδιαίτερα σημαντικά. Και μια τελευταία παρατήρηση. Είναι αδικαιολόγητη αυτή η επιφυλακτικότητα και η διστακτικότητα των ε, εισφορέων των βασικών εισφορέων στον προπολογισμό εδώ ε, πρέπει να ενισχύσουμε την αγορά. Η Ρουμανία έχει χάσει 16.000 γιατρούς και 22.000 μηχανικούς που έχουν μεταναστεύσει σε, στα μεγάλα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συμβάλλουν περισσότερο στον προπολογισμό. Πρέπει λοιπόν να ενισχυθεί πολιτική συνοχή. Ευχαριστούμε κύριος Λόπες Αγγιλάρ. Επίτροπε Χάν, σας υπενθυμίζω ότι ως Επίτροπος που ήσασταν στην περιφερειακή πολιτική, ασχολείστε με την απότερη περιφέρεια, την εξόχως ε, από, από περιφέρεια, θα πρέπει τώρα να δείτε ότι ε, εμείς προερχόμαστε από διαφορετικές πολιτικές ομάδες, αλλά και από τις δύο πλευρές που προερχόμαστε, σοσιαλιστές και δημοκράτες και οι δύο έχουμε την ίδια γραμμή. Ε, τώρα, έχει φτάσει το επίπεδο των παραχών στο πιο τσιγκούνικο επίπεδο της ιστορίας. Ε, είναι απαράδεκτο. Οπότε αυτές οι καινούργιες πολιτικές χρειάζονται, αλλά δεν είναι δυνατόν να γίνονται αυτές οι πολιτικές εις βάρος άλλων πολιτικών, πολιτικής συνοχής, της περιφερειακή πολιτικής, υπέρ των πιο αποκεντρωμένων, των πιο ε, ε, φτωχών περιοχών, εις βάρος της γεωργίας και επίσης και κάτι άλλο, ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει την τελευταία λέξη, αυτό να μην το ξεχάσει κανείς, να μην το αγνοεί κανείς, γιατί εμείς... Ε, ε, πρόκειται να κάνουμε την πλάστη να γύρει για αυτό το δημοσιονομικό πλαίσιο. Οπότε θα πρέπει να κάνετε την αλλαγή, θα πρέπει ε, να κάνετε μια προσαρμογή προς τα απάνω και έτσι να ικανοποιήσετε αυτές τις ανάγκες όπως τα έχει πει το Κοινοβούλιο και τα έχει πει με την ε, ευρύτερη δυνατή πλειοψηφία γιατί η εναλλακτική πάντα είναι το να μπλοκάρουμε, να φρενάρουμε αυτό το δημοσιονομικό πλαίσιο. Αλλιώς πάμε για την χρεοκοπία του ευρωπαϊκού ονείρου. Κυρία Κέλλη. Κύριε Επίτροπε, είναι η ατμομηχανή, είναι ο άξονας της ε, μηχανής του κινητήρα, άρα δεν μπορεί το όχημα να λειτουργήσει χωρίς τον κινητήρα και άρα χωρίς προϋπολογισμό δεν μπορούμε να προχωρήσουμε και όσο πιο ισχυρός ο προπολογισμό, πιο καλά λειτουργεί η Ένωση. Οπότε θα πρέπει το Συμβούλιο και ιδίω οι Πρωθυπουργοί να εξασφαλίσουν ότι ο προπολογισμό να μπορέσει να μας βοηθήσει να κάνουμε αυτό το οποίο ξέρουμε να κάνουμε. Η προστιθέμενη αξία η οικονομίας κλίμακας, ε, γεωργία, συνοχή, κλιματική αλλαγή, έρασμο, έρευνα κλπ. και η απόδοση είναι πολύ μεγάλη, 3-4 ευρώ πολύ για κάθε ευρώ που εμείς εισβάλλουμε. αυτό χρειάζεται να υπάρχει ε, ευρύ πνεύμα, ανοιχτό μυαλό και να αυξηθεί ολονών η συνεισφορά στο, στην υπόθεση αυτή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ε, έγινε κατεξαίρεση αυτό για να δώσω λίγο περισσότερο χρόνο ε, Μια και δεν ήταν ιδιαίτερα φορτωμένη η ημερήσια διάταξη. Οπότε θα ήθελα να δώσω το λόγο τώρα στον κύριο Χάν για να απαντήσει. Uh, Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί ευρωβουλευτέ, σα ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την γόνιμη ανταλλαγή απόψεων. Οι συζητήσει για το επόμενο ε, έχουν τονίσει πόσο μεγάλο πάθος έχουμε όσον αφορά τα θετικά αποτελέσματα και τις επιπτώσεις στους πολίτες μας. Δεν συμφωνούμε σε όλα, όμως υπάρχει συνένεση τουλάχιστον ως προς τις κοινέ μας προτεραιότητες. Ένας προπολογισμό βεβαίως πρέπει να μετουσιωθεί και σε συγκεκριμένους αριθμούς και θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις υψηλές μας ε, προσδοκίες. Ωστόσο, όπως είπε και η πρόεδρος Φοντερ Λάιεν, ο χρόνος μας τελειώνει. Την επόμενη εβδομάδα πρέπει να βρεθεί συμφωνία. Θέλουμε έναν φιλόδοξο προπολογισμό όλοι. Όμως δεν μπορούμε να αγνοήσουμε την πραγματικότητα ότι πλέον είμαστε μια ένωση 27 κρατών μετλών. Και αυτό δημιουργεί προκλήσεις. Και αυτό θα ήθελα να σας καλέσω να επιδιώξουμε έναν προϋπολογισμό ο οποίος να ανταποκρίνεται στους στόχους μας. Και θα χρειαστεί να συνεχίσουμε το έργο μας στις, ε, στους στις τομεακές μας πολιτικές. Και μαζί θα πρέπει να προσπαθήσουμε να αξιοποιήσουμε τον προπολογισμό με τέτοιο τρόπο, ώστε το ευρωπαϊκό θεματολόγιο να εξυπηρετηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Πράσινη συμφωνία για την κλιματική ουδετερότητα και νέοι ήδη πόροι, όπως είναι το, τα πλαστικά και το ETS, για να μπορέσουν να χρηματοδοτηθούν ευρωπαϊκά αγαθά. Επίσης, θέλουμε να γίνουν επικοδομητικές συζητήσεις στη Σύνοδο Κορυφής του, της 20 Φεβρουαρίου για να καταλήξουμε σε ένα καλό αποτέλεσμα για την Ευρώπη. Δεν μπορεί η Ευρώπη να επιτύχει τις προτεραιότητες της και τους στόχους της όταν γίνονται περικοπές εκεί όπου οι πολίτες περιμένουν να γίνουν περισσότερα. Σύνορα, κλίμα, ψηφιοποίηση, εράσμους, άμυνα. Όλα αυτά τα θέματα. Και γι' αυτό δεν έχουμε φτάσει ακόμα στο τέλος των συζητήσεων. Μας τελειώνει ο χρόνος. Έχουμε καθυστερήσει περισσότερο από ότι το 2013, όπου χάθηκε ένα ολόκληρο έτος για πολλά προγράμματα, τα οποία ξεκίνησαν τελικά το 2014. Γι' αυτό θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2021 όλα τα προγράμματα θα έχουν τεθεί σε ισχύ και σε υλοποίηση. Α είμαστε θετικοί, α είμαστε ενωμένοι. Νομίζω ότι το χρωστάμε στου εαυτού μα στα θεσμικά μα όργανα, αλλά κατά κύριο λόγο το οφείλουμε στου πολίτε μα που περιμένουν συγκεκριμένα αποτελέσματα. Η Κομισιόν εκφράζει την προσήλωσή της στον συνεχιζόμενο διάλογο και στην, στις επαφές κατά τη διάρκεια των επικείμενων διαπραγματεύσεων. Και παρεμπιπτόντος, να σας πω ότι έχω ερωτηθεί από πολλούς, ακόμη και σήμερα, αν πιστεύω ότι είναι πιθανό να επιτευχθεί συμφωνία την επόμενη εβδομάδα. Έχοντας κατά νου ότι σύμφωνα με την παράδοση δεν αρκεί μία και μόνο σύνοδο κορυφή για να καταλήξουμε σε συμφωνία. Νομίζω όμω ότι είναι καιρό πια να πάρουμε διαζύγιο από αυτή την παράδοση και να εργαστούμε για μια συμφωνία η οποία θα μπορέσει να επιτευχθεί σε μία και μόνο συνάντηση. Εγώ ταξίδεψα σε πολλά κράτη-μέλη, είχα πολλές συνομιλίες και επαφές τις προηγούμενες εβδομάδες και πιστεύω πραγματικά ότι μπορεί να επιτευχθεί συνένεση μεταξύ των κρατών μελών ακόμη και την επόμενη εβδομάδα υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρξει ε, βούληση, θα υπάρξει δυναμική προς αυτή την κατεύθυνση και με την προϋπόθεση ότι τα μεγάλα ιδίω κράτη-μέλη θα δραστηριοποιηθούν εντονότερα προς την κατεύθυνση της επίτευξης μια συμφωνίας. Γι' αυτό και σας καλώ όλους να ε, ασκήσετε πίεση μέσω των επαφών σας, μέσα από τα, μέσα από τα κόμματά σας, τι ηγεσίε των κομμάτων σας, για να επιτευχθεί μια συμφωνία η οποία θα αποβεί προ όφελο όλων και να μας βοηθήσει να ξεκινήσουμε τις διαπραγματεύσεις με το Κοινοβούλιο. Και εμείς από την πλευρά της Κομισιόν θα κάνουμε ό,τι καλύτερα για να διευκολύνουμε τις διαπραγματεύσεις αυτές. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, Επίτροπη Χάν, και νομίζω καλή δουλειά θα ήταν καλό να συνεχιστεί. Τελευταία, ε, η Υπουργό Γιάνκ. Κυρίε και κύριοι βουλευτές, Κύριε Επιτροπή, σα ευχαριστώ για αυτή την τόσο επικοδομητική συζήτηση. Έχω σημειώσει τι απόψει και ανησυχίε σα και θα φροντίσω να τι μεταφέρω στον Πρόεδρο Μισελ. Είναι σημαντικό η Ευρώπη να συνεχίσει να αναπτύσσεται και τα κοινωνικά και οικονομικά κενά να καλυφθούν. Δηλαδή, οι πολιτικέ που βασίζονται στη συνθήκη να ε, εξακολουθήσουν και να ενισχυθούν. Θα πρέπει όμω να λάβουμε υπόψη και τι νέε προκλήσει που αναφέρονται και στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική Ατζέντα. Επιπλέον, ένα από τα μεγαλύτερα κράτη τη Ευρωπαϊκή Ένωση και απευθεία ε, ε στον προπολογισμό έχει αποχωρήσει. Θα πρέπει λοιπόν να καλύψουμε το κενό στον προπολογισμό και να βεβαιωθούμε ότι έχουμε του πόρου για να επιτύχουμε του στόχου και τι προκλήσει που προκύπτουν από την φιλόδοξη ατζέντα που έχουμε θέσει. Ε, θα πρέπει να ε, καθορίσουμε έναν προπολογισμό ο οποίο να είναι αποτελεσματικό για να καλύψουμε και τους στόχους μας και τις φιλοδοξίες των πολιτών. Σε συνεργασία μαζί σας θέλουμε να βεβαιωθούμε ότι υπάρχει μια ομαλή μετάβαση στον επόμενο δημοσιονομικό κύκλο. Μόλις η αρχική κρατών και κυβερνήσεων στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο φτάνουν σε συμφωνία, η κρατική προεδρία θα είναι έτοιμη να επιταχύνει τι εργασίε για να πετύχει αποτελέσματα και για του πολίτε και για το μέλλον τη Ένωσή μα. Σα ευχαριστώ πολύ και πάλι για την προσοχή σα. Εμείς ευχαριστούμε. Τώρα ολοκληρώνεται η συζήτηση. Θα διακόψουμε μέχρι τις 12. Τότε έχουμε τις ψηφορίες.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 President! Dear colleagues, please take... Καθίστε συνάδελφοι. Θα αρχίσουμε τις ψηφοφορίες. colleagues, could I ask you to take your seats, please? Παρακαλώ, καθίστε ξαναλέει πρόεδρος. Okay. This is the third and last time I will ask you to take your seat. Τρίτη και τελευταία φορά που σας το να καθίσετε πριν αρχίσουμε τις ψηφοφορίες. Of you who are having meetings in the corridors, please take your seats. I am about to start the voting procedure. Αρχίσουμε την ψηφοφορία. Να μην κατονομάσω τους ταραξίες, αλλά θα το κάνω αγρίαστη. Take our seats. Everyone is anxious to get started. Thank you. I just have one announcement to make. Έχω όμως μία ανακοίνωση. Ακούστε παρακαλώ. Το ΕΛΚ μας ειδοποίησε για τις αποφάσεις όσον αφορά την αλλαγή των, του ορισμού των βουλευτών στις επιτροπές. Αυτά θα καταχωρηθούν στα πρακτικά της σημερινής ε, συνόδου και θα έχουν ημερομηνία ε, την ε, ώρα και μέρα της ε, ανακοίνωσης. Ποιος έχει διαδικαστικό πριν την έναρξη της ψηφοφορίας. Ευχαριστώ. Ναι, ναι, διαδικαστικό είναι για τον κανονισμό. Άρθρο 10, παραγράφος 4 ορίζει ότι την ώρα των ε, κοινοβουλευτικών διαδικασιών δεν θα πρέπει να γίνονται ε, υβριστικές διατυπώσεις. Και χθε ο κύριος Μαριάννη, ενώ του κάποια δυσερία, έλεγε ότι θα πρέπει να υποστηρίξουν τον Πασαραπάρ ούτως ώστε να υπάρχει ειρήνη. Και αυτό να γίνει με, με εξόντωση, με εξόντωση των στασιαστών, όχι της ΔΕΣ, όχι να τους καταπολεμήσουμε, όχι να τους πολεμήσουμε, να τους εξοντώσουμε. Αυτό είναι φασισμός, αυτό είναι υβριστικό. Δεν είναι δυνατόν να επιτρέψουμε ε, τους υπηρέτες του Πούτιν να μεταφέρουν εδώ μια τέτοια ανίκια γλώσσα εδώ στο κοινοβούλιο δεν είναι δυνατόν εδώ στο ημικύκλιο να δεχτούμε αυτούς οι οποίοι ε, είναι απολογητές των εγκλημάτων πολέμου. Σύμφωνα με το άρθρο 14 παρακαλώ να επιβληθούν κυρώσεις. Αυτό δεν θα περάσει. Uh, Ο Πρόεδρος, κύριε Γκλίξμαν, ευχαριστούμε που μας επισημάνετε το γεγονός. Θα διαπιστώσουμε από τα πρακτικά τι θα γίνει και θα ειδοποιήσουμε σχετικά τον Πρόεδρο. Έχετε κύριε διαδικαστικό. Παραδόξως, να ευχαριστήσω τον Ραφέλη Γκλουξμαν για τα όσα είπε. Διακόπτεται το μικρόφωνο από την Πρόεδρο. Δεν έχουμε συζήτηση τώρα επί των όσων είπε ο κ. Γκλουξμαν, λέει Πρόεδρος. Θα συνεχίσουμε σύμφωνα με την ημερησία διάταξη. Καλύφθηκε. Ολοκληρώθηκε το θέμα και προχωρούμε. Πρώτα πρώτα, πριν να αρχίσουμε τις ψηφοφορίες. Please have some respect for the chair. Παρακαλώ δείξτε σεβασμό προ την Προεδρία. Ευχαριστώ συναδελφοί και τώρα θα σας διαβάσω μία δήλωση που έχει προκαλέσει την οργή κάποιων συναδέλφων και οπότε θα διαβάσω νυφάλια. Θα πρέπει να σας πενθυμίσω ότι σύμφωνα με την διαδικασία μας ε, πανώ και σημαίες δεν επιτρέπονται. Παρακαλώ οι κλητήρες να καλέσουν τους συναδέλφους να μετακινήσουν σημαίες και πάνω παρακαλώ σεβαστείτε τον κανονισμό λειτουργίας μας όπως προανέφερα. Και τώρα, ψηφοφορίες. Κύριε Λαμπέρ, έχουμε τέσσερις εκθέσεις του κυρίου Μπουρζουά. Ξεκινούμε με την πρώτη που αφορά τη σύναψη ομονίας ελευθέρων συναλλαγών Ευρωπαϊκής Ένωσης Βιετνάμ. Θα γίνει αυτό με ονομαστική ψηφορία. Ψηφίζουμε. And the vote is now closed. Πέρας. Εγκρίνεται. Ψηφοφορία για το ψήφισμα της Συμφωνίας Ελεύθερων Συνελλαγών. Τροπολογία 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 5. Υπέρ.